Καλημέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, νωρίς νωρίς σήμερα. Ξέρω ότι δεν ήθιστε, αλλά βλέπετε έχουμε πολλές ψηφοφορίες και γι' αυτό έπρεπε να αρχίσουμε νωρίς. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Σχόλια παρακαλώ. Όχι. Εγκρίνεται λοιπόν. Συνεχίζουμε. Σημείο 2. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Μία ανακοίνωση έχω να σας κάνω που έχει να κάνει με τη διερμηνία μας σήμερα. Τα σλοβακικά είναι μόνο παθητικά, που σημαίνει ότι μπορείτε να μιλήσετε σλοβακικά αν θέλετε, αλλά δεν μπορείτε να ακούτε σλοβακικά. Τις άλλες γλώσσες τις έχουμε. Σημείο 3 πρώτη μας ψηφοφορία, αλλά πριν ψηφίσουμε να καλωσορίσω εδώ σήμερα μια ομάδα επισκεπτών ιδιαίτερη. Είμαι από την Βόρεια Γερμανία, όπως ξέρετε, από το Κουκστάντερ που είναι στη Βόρεια Γερμανία και με, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα σήμερα που καλωσορίζω εδώ μια αντιπροσωπεία στρατιωτικών αντρών και γυναικών από την Τέριγα 3, που είναι μια γερμανική στρατιωτική μονάδα. Όλοι αυτοί οι στρατιώτες έχουν συμμετάσχει στο κέρας της Αφρικής σε ευρωπαϊκές αποστολές. Καλώς ήρθατε. Okay. Καλώς. Συνεχίζουμε λοιπόν και ψηφίζουμε έκθεση σχετικά με την έκθεση Επιτροπής του 2018 για την Βοσνία Ζεγοβίνη. Ο Κριστιαν Νταν Πρέντα είναι ο εισηγητής μας. Παρακαλώ. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Χαίρομαι που θα ψηφίσουμε σήμερα το πρωί αυτή την έκθεση της Επιτροπής για τη Βοσνία Ζεγοβίνη και θέλω να ζητήσω στην Ολομέλεια να μην έχουμε αυτή την έκθεση στην ημερήσια διάταξη πριν να εγκρίνει τους διαδικαστικούς κανόνες το Κοινοβούλιο της Βοσνίας Ζαγοβίνης. Ακόμα δεν έχει ψηφίσει περιμένουμε να δημιουργηθεί ο μηχανισμός στη Βοσνία Ζεγοβίνη, οπότε πιστεύουμε ότι πρέπει να αναβληθεί η ψηφοφορία, ώστε προηγουμένω να μα πάρει στα σοβαρά το Κοινοβούλιο της Βοσνίας Ζεγοβίνης. Συνεπώ, να μην ψηφιστεί η έκθεση αυτή, παρά μόνο αφού η Βοσνία Ζεγοβίνη δείξει ότι όντω θέλει να έρθει προ εμά. Κριστιαν Πρέντα, λες να μην ψηφίσουμε σήμερα. Ναι, στην Επιτροπή μας να ψηφίσουμε, στην Ολομέλεια να μην ψηφίσουμε. Να μην στείλουμε δηλαδή την έκθεση αυτή στην Ολομέλεια, αλλά να περιμένουμε πρώτα να εγκρίνουν τους διαδικαστικούς κανόνες στη Βοσνία Ριζεγοβίνη πρώτα. Ωραία, άλλα σχόλια έχει κανείς κάτι να πει. Όχι από ό,τι βλέπω. Καλώς. Αρχίζουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Μπορείτε να ψηφίσετε. Α, απορρίφθηκε. Συμβαστική 3 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 53 με ονομαστική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίφθηκε 20 κατά 19 υπέρ. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 64 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ψηφίστε παρακαλώ. Άλλος ένας πρέπει να ψηφίσει. Εγκρίθηκε. 21-19. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 111. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Όλα τσίμα τσίμα οι με το πριν 12 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 138 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 159 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 159 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 21 υπέρ,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 Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 19. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε, σαφώς. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Φετολικές αναφορέ 1 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ, όχι, η 7 καταπίπτει. Προφορική 2 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά αποχές. Θα ελέγξουμε την 8 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. 9 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Τελική ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία. Η εννέα απορρίφθηκε. Τέλος, εγκρίθηκε 33 ψήφοι υπέρ, 7 κατά και 2 αποχές. Και περνάμε στο σημείο 4, πρωτόκολλο τη Συμφωνία για τη Σύναψη Εταιρική Σχέση και Συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών του αφενό και τη Δημοκρατία του Κυργιστάν αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση τη Δημοκρατία τη Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκητή μα είναι, τι έκπληξη, ο κύριο Ντεν Πρέντα. Θέλετε το λόγο, κύριε Ντεν Πρέντα. Όχι. Καλώ Έχουμε μία ψηφοφορία όλοι και όλοι. Η ηλεκτρονική για το σχέδιο αυτό. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Και εγκρίθηκε. 40 υπέρ, μία ψήφος κατά. Περνάμε τώρα στο ψήφισμα. Ε, σύσταση προς το Συμβούλιο Επιτροπή και Αντιπρόεδρο Επιτροπής είπε ότι εκπρόσωπο Ένωσης ε, ε, σχετικά με τη Συντολική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κυργυζία. Θέλετε κύριε Πρέντα ο να πάρετε το λόγο. Ψηφίζουμε. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 7 υπέρ κατά ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία υπαριθμών 7. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 37. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές. Άρχεται η ψηφοφορία, η ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 18 του κυρίου Σόλτς. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 του κυρίου Σόλτς υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 33 υπέρ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 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία πάει 79. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και επομένως τώρα θα ψηφίσουμε για την τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για την τροποποιημένη λοιπόν έκθεση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Και εγκρίνεται 40 ψήφοι υπέρ, μία κατά δύο αποχές. Φτάνουμε στο σημείο 6 της ημερησίας διατάξεως. Κατευθυντήριες γραμμές Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντολή του Ειδικού Επεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας πεπιθήσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εισηγητή ο Αντρέι Γκριμπ. Κύριε συνάδελφε, θέλετε να πάρετε το λόγο. Α, δεν είναι καν εδώ. Επομένω, πώ θα πάρετε το λόγο, λέει ο πρόεδρο. Πρόκειται για έναν πολύ μακροσκελή κατάλογο ψηφοφορία. Ξεκινούμε. Συμβιβαστική 1. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 2. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 71. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Η 72 καταπίπτει, συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 81 της κυρίας Βερζιά, άρχεται η ψηφοφορία. 21 προς 21, επομένως απορρίπτεται η τροπολογία 81. Τροπολογία 82 υπέρ κατά αποχές. Θα ήθελα να κάνουμε ηλεκτρονική παλήθευση και για την τροπολογία 82 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Επίσης ε, απορρίπτεται με την ίδια ε, σχέση ψήφων συμβαστική 4 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 5 ομοίως, συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 98, γκριμπ, υπέρ κατά εγκρίνεται. Α, θέλετε να ελέγξουμε την τροπολογία αυτή. 98, επαληθεύουμε ηλεκτρονικά, πέρα της ψηφοφορίας, ε, εγκρίνεται σαφέστατα 31-11, συμβαστική 7 υπερκατά εγκρίνεται, τροπολογία 104 υπερκατά εγκρίνεται.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 Τροπολογία 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. 163 ε, ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και σαφώς απορρίπτεται. Τροπολογία 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 164. 164 Α, πρώτη φορά θα παίρναγε τροπολογία του κυρίου Σουαπχάουζερ. 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 165. Απερίφθη 164 και επομένω πρέπει να ψηφίσουμε την 165. Υπέρ, κατά, αποχέσε, η ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 165.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 Έκθεση, ε, συγγνώμη, τροπολογία Σαφχάουζερ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση, ναι, να επαληθεύσουμε για την τροπολογία 191. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 43 ε, ψήφοι κατά, μία ψήφος υπέρ. Τροπολογία 192 υπέρ κατά αποχές. Θα ε, κάνουμε την επαλήθευση ηλεκτρονική για την τροπολογία 192 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 210 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 210 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να υπαλληθεύσουμε τροπολογία 15, άρχια διαψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18. So we'd have to 18 in favor. Άρα να ψηφίσουμε και τη 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση όπως θέλετε. Για την τροπολογία 18 λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Το είδα, Κρίστιαν, αυτό που λες. Συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 του κυρίου Χάν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 του κυρίου Μισελ υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 31 Μισελ. Πέρας και εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές Προτιμώ να ελέγξουμε. Τροπολογία 42 της κυρίας Βερζιά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45... Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 44 υπέρ. Ε, συγγνώμη, πέρα στις πληροφορίες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές και εδώ να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για τροπολογία 45 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και επίσης εγκρίνεται. Η 46 καταπίπτει. Ε, Αιτιολογικέ αναφορέ τώρα. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 3 δεν ψηφίζεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Α, ε, θα ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 5. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές. Ε, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 6. Ψηφίζουμε. Πέρας και απερίφθη επίση η τροπολογία 6. Η τροπολογία 7 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 8 τη Σβερζιά, Βερζιά υπέρ κατά αποχέ. Η ηλεκτρονική επαλήθευση τη τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 9 σολέ υπέρ κατά κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ερχόμαστε πλέον στην τελική ψηφοφορία όσο ε, ε, επί του ψηφίσματος άρχεται η ψηφοφορία πέρασε και εγκρίνεται 41 ψήφοι υπέρ, 1 κατά, δύο αποχές. Και περνάμε στο σημείο 7, θέσπιση Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης. Συντάκτης της γνωμοδότησης είναι ο αντιπρόεδρός μας, ο κύριος Βίστισεν. Άντερς, θέλεις το λόγο? Πού είσαι? Α, να είσαι. Όχι. I'm supposed to inform colleagues. Λοιπόν, πρέπει να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι αν εγκριθεί η τροπολογία 125, καταπίπτει η τροπολογία 126. Πάμε λοιπόν στην πληροφορία επί της ε, γνωμοδότησης αυτής. Είναι μακρά η ψηφοφορία αυτή. Πολύ μεγάλος κατάλογος ψηφοφορίας. Για γνωμοδότηση όλα τι να πω. Λοιπόν, 10 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε. Ψηφίζεται. τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 77 in favor. 77 υπέρ. Κατά απόχέ. Ωραία θα περάσουμε. Πάμε ξανά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Here, four colleagues are not on board. Λοιπόν, τέσσερις δεν έχουν ψηφίσει. Εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε. Close. Πέρας, απερίφθη. 79 της κυρίας Βερζιά, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Τροπολογία 83 ψηφίζεται παρακαλώ. Πέρας απορρίπτεται. 84 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Τέλεια, πάμε στην 90 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές, ελέγχουμε. Ψηφίζεται επί 91 ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεν ξέρουμε οπότε ελέγχουμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 92 Λόπεζ πέρας της φεφορίας εγκρίνεται μεγάλη διαφορά 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 95 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά αποχές ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 96. It's closed. Πέραση ψηφοφορίας απορρίφθηκε. 97 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 4. 4. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 100 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 100. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Ψηφίζετε σας παρακαλώ επιστροπολογίες 112 ηλεκτρονικά με τις συσκευές σας. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. 5 του κυρίου Βίστησεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ή να το ελέγξουμε καλύτερα. Το ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί τη τροπολογία αυτή. Ψηφίζετε παρακαλώ. Πέρας τη ψηφοφορία, εγκρίθηκε. Γεια σας και θα τα πούμε αργότερα. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 117. Πέρα της ψηφοφορίας. Πολύ κοντά. Εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά You don't δεν έχω το σωστό κατάλογο ψηφοφορίας, μάλιστα. Μόλις με ενημερώνουν από το κοντρόλ. Δεν ψηφίζουμε επί της έκθεσης για το Τατζικιστάν, σωστά. Λοιπόν, ο κατάλογος ψηφοφορία που είχε στη διάθεση του ΕΛΚ είναι εσφαλμένος. Πάμε στο 124. Κυρία Μούντι, σωστά. Τα λέω. Ωραία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Ψηφίζετε σας παρακαλώ ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 124. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Α, και τώρα έρχεται η διαβόητη 125. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Επαλήθευση. Ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 125. Της κυρίας Βερζιά. The vote is closed. Πέρας. Απερίφθη με μεγάλη διαφορά. Και τώρα πάμε στην 126. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα την ελέγξουμε και αυτήν. Ψηφίζετε σας παρακαλώ ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 126. Άρχεται η ψηφοφορία. Μπορώ να επιστρέψω εγώ στο δικό μου κατάλογο τώρα ή όχι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Ωραία. Πάμε στην 127. Περ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Ψηφίζουμε επί της 127. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορία, Εγκρίθηκε. Πού πήγε τώρα ο κατάλογος της ψηφοφορίας μου. Okay, I don't care. Here? So, 127, that was a... 127 είπαμε εγκρίθηκε, σωστά, ωραία, πάμε. 128 υπέρ κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 129 υπέρ κατά, αποχές, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας, απερίφθη. 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ 134 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρα, vote Πέρας. Απερίφημη μεγάλη διαφορά. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 136 τη κύρια Μούντι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 137 υπέρ κατά αποχές Α το ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί τη 137. Σα παρακαλώ, ψηφίζετε. Πέρας τη ψηφοφορία. απερίφθη. 138 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 139 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ψηφίζετε σας παρακαλώ επί της τροπολογίας 139 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία Πέρα της ψηφοφορίας απερίφθη 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6, 7, 8 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 144 έως 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 145, 147, 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 143, 148, 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Όχι, καλύτερα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για την τελευταία ψηφοφορία, 143, 148, 150 Ψηφίζετε. Α, εγκρίνονται. Μπράβο σας. Έχετε εξαιρετική όραση, βλέπω. 152 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 153 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 154 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 157 ε, υπέρ κατά αποχές Ας το ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίζετε σας παρακαλώ επί της 157. Απερίφθη. 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ, κατά αποχές Ας το ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της 162. Ψηφίζετε σας παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη. 163 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 165 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. Ελέγχουμε. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της 165. Άρχεται η ψηφοφορία. It's Πέρας. Απερίφθη. 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ του κυρίου Βίσισεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ...169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. 170 ψηφίζεται.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 κατά αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Όχι, ας το ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίζουμε επί 180 ηλεκτρονικά πέρα της ψηφοφορίας απερίφθη. 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. 2 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ της κυρίας Βερζιά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Ψηφίζουμε επί της 18 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 19 του κυρίου Επιτίδιου. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 31 Βερζιά υπέρ κατά αποχές. Ας το ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 31 της κυρίας Βερζιά. Πολλές αποχές είδα. Πέρασε. Απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Να την ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 36 της κυρίας Βερζιά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Κυρία Πόστ, υπέρ. Ε, τότε εγκρίνεται. Τίποτα, τίποτα, μην ανησυχείτε. Έριξα απλά τον καφέ μου. Δεν έχει σχέση με την ψηφοφορία. Λοιπόν, πού πάμε. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές το ελέγχουμε. Ψηφίζουμε επί της τροπολογίας 39 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθημη μεγάλη διαφορά. 40 επιτίδιος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε τροπολογία 41 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά σας παρακαλώ επί τη τροπολογία 41 τη κυρία Βερζιά πέρα της ψηφοφορίας απερίφθη 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 Καστάλντο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επιστροπολογία 47 πέρας της ψηφοφορίας. Κυρία Πόστ, εσείς υπέρ, άρα εγκρίνετε. 48 κατά πίπτη, 49 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά αποχές Απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές Ας ψηφίσουμε καλύτερα χρονικά επιστροπολογίες 54. Ψηφίστε σας παρακαλώ. Κυρία Πόστ, εσείς αποφασίζετε πού θα γύρει πλάστιγκα σήμερα υπέρ λοιπόν, άρα η τροπολογία αυτή εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 3 καταπίπτει, το ίδιο και 57, το ίδιο και 58, οπότε πάμε βερζιά 59 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται.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 66 του κυρίου Ράιμον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της 65 της κυρίας Βερζιά πέρας της ψηφοφορίας. Και χάρη στην κυρία Πόστ εγκρίνεται. 67 Καταπίπτει. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν καταπίπτει. Ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε. Ψηφίζουμε επί 72, άρχεται ψηφοφορία. πέρας, απερίφθη, 73 υπέρ κατά αποχές, θα ελέγξουμε, ψηφίστε σας παρακαλώ, επί της τροπολογίας αυτής, πέρας, απερίφθη, 74 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές αναφορές 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του σχεδίου γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζετε σας παρακαλώ. The τη is και απερίφθη με 19 ψήφους υπέρ, 24 κατά. Mr. Brock. Κύριε, Κύριε Μπροκ, παρακαλώ. Θέλω να ετυλογήσω την ε, ψήφο μου. Εγώ είμαι υπέρ του Ταμείου που σχεδιάζεται, αλλά θα ήθελα να είχαν γίνει περισσότερες διαβουλεύσεις, να είχαμε βρει περισσότερους συμβασμούς. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό και γι' αυτό καταψηφίσαμε ε, την γνωμοδότηση. Η ψήφος μας αυτή δεν στρέφεται κατά του Ταμείου, αυτού καθ' αυτού, αλλά ε, ε, ε κατά της διαδικασίας που ακολουθήθηκε εδώ στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλουν άλλοι συνάδελφοι το λόγο. Κυρία Επιτίδιε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι η ψήφος αυτή είναι εναντίον του Ταμείου, διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες και λαοί οι οποίοι να υποφέρουν οικονομικά όπως ο ελληνικός λαός και εμείς να διαθέτουμε χρήματα για τους παράνομους μετανάστες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πετιδίου. Άλλος κανείς. Νελίτς, ναι, ναι, παρακαλώ. Ε, απορρίπτω πλήρως ε, αυτή την τελευταία τοποθέτηση. Δυστυχώς λυπάμαι και εγώ για το γεγονός ότι δεν ε, ε κατέστη δυνατόν να βρεθούν συμβιβασμοί. Δεν ξέρω πώ μπορούμε να ακολουθήσουμε μια διαφορετική διαδικασία. Πάντω είναι πολύ αρνητικό το μήνυμα αυτό που στέλνουμε σήμερα ω Κοινοβούλιο. Το γεγονό δηλαδή ότι απερίφθη αυτή η γνωμοδότηση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Οστρεβίτσιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι μια δήλωση της ΑΛΤΑ. Εμείς υπερψηφίσαμε το ταμείο αυτό χάσαμε. Δεν μας άρεσε ο τρόπος με τον οποίο διατυπώθηκε αυτή η γνωμοδότηση. Δεν έγιναν σχεδόν καθόλου διαβουλεύσεις. Το ΕΛΚ, οι σοσιαλιστές, εμείς είχαμε μια κοινή γνωμοδότηση για κάποιες συμβαστικές προτάσεις, αλλά δεν ήταν αρκετό. Αν είχε εγκριθεί η γνωμοδότηση που θα διέγραφε το επεξηγηματικό κομμάτι. Ήμασταν κατά, έτσι καλώς δεν έγινε, χάσαμε την ψηφοφορία. Χρειάζεται όμως το ταμείο αυτό. Ο τρόπος που ψηφίσαμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι ατυχές. Πρόεδρος, έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ τα πράγματα δεν εγκρίθηκε η γνωμοδότηση που σημαίνει ότι εμείς ε, δεν θα δώσουμε την γνωμοδότησή μας Τώρα για τροπολογίες στη Λίμπε, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, πάντως στη Λίμπε πρέπει να υποβάλουμε τροπολογίες αν θέλουμε κάτι να κάνουμε εδώ. Τελείωσε. Ό,τι είχαμε να κάνουμε εδώ το κάναμε, τελειώσαμε. Πότε ψηφίζει Λίμπε? «11 Δεκεμβρίου προθεσμία για τροπολογία στη Λίμπε». Καλώς το ξέρετε συνάδελφοι. Οπότε περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία, το σημείο 8. Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων στα πλαίσια του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Η συγητής είναι ο Έντουαρτ Κούκαν. Παρακαλώ. Να ψηφίσουμε. Εξαιρετική γνωμοδότηση αυτή. πρώτες ψηφοφορίες. 64 με 160 ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε για την 44. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Η κυρία Πώστα έφυγε. Τι έγινε. Δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. 45. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται νομίζω, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. 47. Τέλος. Εγκρίθηκε. Καταπίπτει 48. 49 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε για την 50. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. 52 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ.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 κατά, αποχές, απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 63. Ψηφίστε. Τέλος, απορρίφθηκε. Κυρία Βερζιά, πολλή δουλειά έχετε. 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά, Αποχέ, απορρίπτεται. 77 υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 80. Τέλος, απορρίφθηκε σαφώς. 81 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε 82 ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε. 83 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θα ελέγξουμε. 88. Ψηφίστε παρακαλώ. Εγκρίθηκε. 89 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κύριε Κούκαν, 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε την 108. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Απορρίφθηκε. 109 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε 111. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Απορρίφθηκε. 113 υπέρ,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 Φύτε 129 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. 129. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άλλοι τρεις. Απορρίφθηκε. 130 υπέρ, κατά αποχές. Οι φιλελεύθεροι τι λένε, 130 Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 131 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε. 131. Τέλος. Απορρίφθηκε σαφώ. 132 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ, κατά αποχές 135 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 135 να ελέγξουμε, καλώς. Απορρίφθηκε. 136 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 137 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 138 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 139 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 142 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ,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 κατά, αποχές, απορρίπτεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και φτάνουμε στις ετουλογικές σκέψεις. 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε για την 7. Ψηφίστε παρακαλώ. Φύτο, 7. Τέλος, απορρίφθηκε πραγματικά. 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε 10. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Τέλος, απορρίφθηκε. 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά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 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 36 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 36 άρχεται η ψηφοφορία. <clears throat> Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, υπαριθμόν 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39. Α, 38 ηλεκτρονική επαλήθευση βεβαίως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ο Έλμαρ έφυγε. <clears throat> Επομένως, τροπολογία 39 της κυρίας Βερζιά, υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Ε, τώρα θέλεις, έχουμε δύο ακόμα τροπολογίες να ψηφίσουμε. Κύριε Πρέντα, παρακαλώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Βερζιά γιατί έχει υποβάλει 113 τροπολογίες. Είναι ρεκόρ ακόμα για την Επιτροπή μας. Την ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία ε, Βερζιά λέει χαίρομαι πάρα πολύ όταν με συγχαίρει ο κύριος Πρέντα. Εδώ ξεκινάει λοιπόν μια καινούργια φιλία, λέει ο πρόεδρος. Ε, την 43 την ψηφίσαμε, όχι. Την ψηφίσαμε, ρωτάει ο πρόεδρος. Έχουμε τώρα μόνο την τροπολογία 4 του κυρίου Φρουνζουλίκα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και ε, διανομαστικής κλίσεως το τροποποιημένο κείμενο. Ψηφίζουμε. Πέρασε και εγκρίνεται 32 ψήφοι υπέρ 4 κατά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι ε, και τώρα θα δώσω τον, ε, την Προεδρία στον κύριο Φρόντ. Σε τρία λεπτά θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Good Καλημέρα και πάλι και από μένα. Δεν είναι η πρώτη φορά που προεδρεύω, αλλά χαίρομαι τόσο πολύ που είναι σαν να είναι η πρώτη φορά. Ναι, κύριε Πρέντα, τώρα εμένα θα έχετε απέναντί σας. Τι να κάνετε για καμιά ώρα. Συνεχίζουμε λοιπόν με μία έκθεση η οποία αφορά τη σχέση με το Τουρκμενιστάν και θα δώσω το λόγο στην κυρία Μανέσκου. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Μανέσκου. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ε, καλωσορίσω τη θέση της κυρίας ε, Μογκερίνη που στέλνει αντιπροσωπεία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τουρκμενιστάν. Είναι μια προσπάθεια η οποία εν τέλει στέφεται από επιτυχία. Θα πρέπει βεβαίω να δείξουμε και εμείς, όπως έχω πει και επανειλημμένα, ότι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εμπλακεί πλήρω ε, σε συμφωνία εταιρική σχέση με το Τουρκμενιστάν που θα περιλαμβάνει και το, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το εμπόριο. Ε, τομεακός διάλογο και συνεργασία λοιπόν με το Τουρκμενιστάν. Στο κείμενο που προτείνεται το ψήφισμα ε, ε, αναφέρει ε, ότι ε, πριν δώσουμε την συνένεσή μας θα πρέπει οπωσδήποτε να περιληφθούν τα, τα, τα ε, ε, κατωτέρω στοιχεία συστάσεις ε, βράχη πρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες όταν αφορά την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διακυβέρνηση και ε, δημόσιε ε, δεσμεύσεις όσον αφορά τους μηχανισμούς παρακολούθησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων που προτείνει η κυρία Μογκερίνη. Ελπίζω ότι θα βρούμε εντελή πολιτικά κοινό τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά από όλε τι πολιτικέ ομάδε, ε, γιατί με τον τρόπο αυτό θα καθορίσουμε καλύτερα τι μελλοντικέ σχέσει μα με το Τουρμενιστάν. Θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα κατά περιόδους να αξιολογούμε ε, και να έχουμε επισκόπηση και αναφορά των, ε, της πρόοδου. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους και από τους σκιώδεις εισηγητές να στείλουν τις τροπολογίες τους και σας ε, ε, βεβαιώ ότι από τη δική μου πλευρά είμαι διατεθειμένη να συνεργαστούμε καλά έτσι ώστε το κείμενο να είναι αποτελεσματικό και σωστό στο τέλος. 11 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί λίγη η προθεσμία υποβολής των τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μανέσκου και εγώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ε, λόγω της ε, μακράς ψηφοφορίας δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα πρέπει να τελειώσουμε μέχρι τις 10 ε, και έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην κοινή μας συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Ο κύριος Άλλη θέλει να μιλήσει. Δύο λεπτάκια παρακαλώ, όχι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σκιώδηση της για την Άλντε. Κυρία Μανέσκου, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια ε, για την ενδιάμεση έκθεση, η οποία ε, με ισορροπημένο τρόπο ε, παρουσιάζει τις σχέσεις μας με το Τουρκμενιστάν. Εκτιμούμε θετικά την αναφορά σε βράχη πρόθεσμα benchmarks, καθώς επίσης και την ανάγκη υποβολής ενδιαμέσων εκθέσεων. Θέλουμε πάντως κάποιες εξηγήσεις. Ανθρώπινα δικαιώματα βήματα ε, βήματα απαραίτητα ε, ε, έτσι ώστε να ληφθούν, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οπωσδήποτε στην εταιρική σχέση συνεργασίας. Για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται και αναθεώρηση του συντάγματος καθώς επίσης και βελτίωση των, της ε, υλοποίηση των όσων ε, η Βουλή του Τουρκμενιστάν έχει ε, ψηφίσει. Επίσης, διαβούλευση με διεθνείς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σχετικά με την συμμόρφωση του Τουρκμενιστάν προς τις βασικές δημοκρατικές αρχές. Επίσης, όλα τα στοιχεία τα οποία θεσμοθετούν την πλουραλιστική πολυφωνική δημοκρατία. Άλλο στοιχείο είναι ότι δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το θέμα της ε, επιτήρησης monitoring από διεθνείς ανεξάρτητους οργανισμούς της κατάστασης ε, στο Τουρκμενιστάν. Επίσης, ε, το 2017 έγινε μια αποστολή εμπειρογνωμόνων ε, στο Τουρκμενιστάν. Θα πρέπει να επιτρέψει το Τουρκμενιστάν και άλλες ε, παρόμοιες αποστολές. Θα πρέπει επίσης το Τουρκμενιστάν να ενεργήσει έτσι ώστε να καταπολεμηθούν τρομοκρατία, διασυνοριακή εγκληματικότητα, λαθρεμπόριο ναρκωτικών ουσιών κλπ. και ε, αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ε, προώθησης ε, από το Τουρκμενιστάν του περιφερειακού διαλόγου. Τέλος, υλοποίηση και θέσπιση των δημοκρατικών αρχών και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στοιχεία εκ των Ουκάνεφ για την Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπόρις Γιαλότσεβιτς από την Εξωτερική Υπηρεσία την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζουμε βεβαίω την έκθεση. Πράγματι, η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος, η κυρία Μογκερίνη, ανακοίνωσε την αποστολή ε, μιας αντιπροσωπείας το 2019 που θα μας επιτρέψει να παρακολουθήσουμε στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα να υπάρχει ένας πιο άμεσος διάλογος με την κυβέρνηση της χώρας και να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή των διαφόρων συμφωνιών που έχουμε συνάψει με το Τουρκμενιστάν. Βεβαίως πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Οι αλλαγές ε, δεν, μπορούν, ε, δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα γίνουν εν μία νυχτά. Είναι μεγάλη η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, παρόμοια με εκείνη που ακολουθείται και με το Ουσμπεκιστάν. Παρ' όλα αυτά αποτελούν μια θετική βάση για καλές σχέσεις, οι οποίες θα ε, παρακολουθούν και θα συνοδεύουν πάντοτε τις μεταρρυθμίσεις, καθώς αυτές θα υλοποιούνται και θα μεταρρυθμίζονται. Βεβαίως, θέλω επίσης να επισημάνω τον θετικό ρόλο που διαδραματίζει το Τουρκμενιστάν στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας. Είχαμε πριν από 10 μέρες μια υπουργική συνδιάσκεψη, ε, στην οποία παρέστη το Τουρκμενιστάν και εκεί απέδειξε ότι πραγματικά μπορεί να παίξει ηγετικό ρόλο, ε, ιδίω όσον αφορά την διαχείριση των υδάτων με το Ταμείο της Αράλης. Χαιρετίζουμε την έκθεση λοιπόν, αλλά υπενθυμίζω ότι πραγματικά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όσον αφορά τα όσα μπορούν να επιτευχθούν βραχυπρόθεσμα από την χώρα αυτή, το Τουρκμενιστάν. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να σα υπενθυμίσω ότι η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων θα γίνει στι 21 Ιανουαρίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει στι 4 Φεβρουαρίου. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει στην ε, πρώτη ε, Σύνοδο Ολομέλειας ε, του Μαρτίου του 2019. Περνάμε στο επόμενο σημείο της τη διάταξη, Κατάσταση των πολιτικών σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία. Θα συζητήσουμε το σχέδιο έκθεση που έχει συντάξει η κυρία Καλνιέτε. Όπως γνωρίζετε, οι σχέσεις με τη Ρωσία ήταν δύσκολες τα τελευταία χρόνια. Ιδίως λόγω του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία, την κατοχή της Κρυμαίας και τις συζητήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή της Συμφωνίας του Μίνσκ. Την προηγούμενη εβδομάδα Είδαμε και μια κλιμάκωση της κατάστασης στην Αζωφική θάλασσα που οδήγησαν στα γεγονότα που εμείς καταδικάσαμε ε, εδώ στο Κοινοβούλιο. Θέλουμε η Ρωσία να ε, αποκαταστήσει την πλήρη ελευθερία στα στενά του Κέρτς. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερα χρόνια από την ε, έγκριση της έκθεσης Λάνσμπερι για την κατάσταση των πολιτικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Και πρέπει δυστυχώς να πω ότι η κατάσταση σήμερα των σχέσεών μας είναι χειρότερη από ό,τι ήταν το 2015. Από το 2015 και την σχετική έκθεση η Ρωσία έχει καταστροφικά ε, παρέμβει στη Σωρία υποστηρίζοντα τον Ασάντ έχει ενισχύσει τις στρατιωτικές της θέσεις, έχει υπογράψει ε, μεγάλες στρατιωτικές συμφωνίες, έχει παραβιάσει συμφωνίες για τον έλεγχο των οπλικών συστημάτων και την συνθήκη του ΖΑΕΒ. Έχει ξεκινήσει επιθέσεις στον κυβερνοχώρο για να ε, εντείνει τις, ε, τις ταραχές ή και για να παρέμβει σε εκλογικές διαδικασίες στην Ευρώπη. Έχει επίσης ε, χρησιμοποιήσει ε, έχει υποστηρίξει ε, επίσης χημικές επιθέσεις στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, επίσης φυλακίζει τους αντιφρονούντες στο έδαφος της. Δεν υπάρχει καμία πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκ. η Μόσχα υποστήριξε τις παράνομες εκλογές στον Ντομπάς και είδαμε και τις τελευταίες ε, εξελίξεις στην Αζωφική θάλασσα. Δυστυχώς όλα αυτά μας οδηγούν σε μια αρνητική αξιολόγηση των σχέσεων μας. Στην έκθεσή μου καλό να γίνουν διάφορα πράγματα. Μη συνέχιση της εθερικής ε, σχέσης και της συμφωνίας ε, συνεργασίας με τη Ρωσία που έτσι και αλλιώς είναι πλέον παροχημένη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγκρίνει περισσότερες κυρώσεις και ατομικά στοχευμένες. Θα πρέπει να, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαγορεύσει πλήρως τις θεωρήσεις και να παγώσει ε, εκείνους που εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να σταματήσει έργα που δεν συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενέργεια και την Ασφάλεια. Τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη θα πρέπει να, να διακόψουν τα προγράμματα χρυσή βίζας που δίνουν και να ενισχυθεί ο συντονισμός και η συνεργασία προκειμένου να ε, ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές αξίες στη ρωσική γλώσσα. Βεβαίως, πιστεύω ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν τον ε, Μάρτιο του 2016 στο Συμβούλιο ε, Ασφαλείας πρέπει να συνεχιστούν, να εφαρμόζονται πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας σε τομεί όπω η κλιματική αλλαγή, η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και η καταπολέμηση τη τρομοκρατίας. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τρόπους για την αποκλιμάκωση των εντάσεων που υπάρχουν μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας και να ε, προσδιορίσουμε μέτρα για την αποφυγή ε, εσφαλμένων εκτιμήσεων και παρανοήσεων. Γι' αυτό θέλουμε να καλέσουμε την ε, Ρωσία να ε, ε, προσέλθει σε συζητήσεις για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνη στο Ντόν και στην Αζωφική θάλασσα. Προσπαθούμε πλέον να αποφύγουμε την κλιμάκωση στρατιωτικών ή κυβερνοεντάσεων και όχι στη φάση οικοδόμησης ε, σχέσεων εμπιστοσύνης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε χώρο ούτε δυναμική για να ξεκινήσει μια νέα πρωτοβουλία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποσυνδεθούμε, να αποσυνδεθούμε πλήρως. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, τις ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκών και να συνεχίσουμε την υποστήριξή μας σε ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, ε, την ελευθερία των δημοσιογράφων. Πρέπει δυστυχώς να ξυπνήσουμε. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βρίσκεται στον, ε, στο μέσο μιας διαμάχης ανάμεσα στη δημοκρατία που βασίζεται σε νόμους και τον αυταρχισμό. Θέλω να έχουμε μια γόνιμη συζήτηση και επικοδομητικές συνεισφορές στην σχέδια έκθεσης, στο σχέδιο έκθεσης. Προθεσμία 10 Ιανουαρίου 10 το πρωί. Και ολοκληρώνοντας θέλω να πω ότι πολύ σπάνια παίρνω το λόγο εδώ στην Επιτροπή. Γι' αυτό και ε, ήθελα να παρουσιάσω εκτενώς την έκθεσή μου αυτή. Ευχαριστώ κυρία Καλνιέτε. Εγώ θα μιλήσω εκ μέρους του, της κυρίας Γιακονσάρη που ζητά συγγνώμη που δεν κατάφερε να παραστεί σήμερα εδώ. Αλλά είναι η εκατοστή πρώτη επέτειος της ανεξαρτησίας της Φιλανδίας. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ. Εκ μέρους λοιπόν της κυρίας Γιακονσάρη θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της και θα συμφωνήσω κι εγώ ότι υπάρχει πολύ χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και στις δύο πλευρές. Το status quo των σχέσεών μας ε, αντιμετωπίζει αδιέξοδα και προκλήσεις. Είναι ατυχές το γεγονός ότι οι συμφωνίες του Μίνσκ δεν έχουν εφαρμοστεί και ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Αναμφισβήτητα είναι σαφές ότι οι σχέσεις μας με τη Ρωσία πρέπει να βασίζονται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε, είναι σοφό να συνεχίσουμε την επικοδομητική συνεργασία σε εκείνους τομείς όπου αυτό είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, στην ε, εταιρική σχέση της Βόρειας Διάστασης, στον, ε, στη συνεργασία στην Αρκτική, στο Μπάρεντς, ε, είναι σημαντικό επίσης να υποστηρίξουμε, από τη Ρωσία, τη συμφωνία με το Ιράν. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι για την αποκλιμάκωση της έντασης και στο πλαίσιο αυτό θεωρώ ότι οι διαβουλεύσεις με τους βουλευτές της Ρωσίας θα ήταν πολύ σημαντικό στοιχείο. Γι' αυτό είναι σημαντικό και οι δύο πλευρές να άρουν τα εμπόδια ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν και πάλι διακοινοβουλευτικές συνδεθκέψεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τη δυναμική που υπάρχει σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα η ψηφιοποίηση, ιδίως όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και την ρομποτική. Και μια τελευταία παρατήρηση. Στον μεγάλο κατάλογο των προκλήσεων και των αδιεξόδων δεν υπάρχουν δύο ε, στοιχεία. Η υποστήριξη της Ρωσίας στην ακροδεξιά στην Ευρώπη και οι εξτρατείες παραπληροφόρησης. Αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το να προσπαθεί κανείς μέσω ψευδών ειδήσεων να παραπλανήσει την κοινή γνώμη είναι ε, μια στάση απαράδεκτη. Δυστυχώς βλέπουμε όμως να συμβαίνουν τέτοια πράγματα και στις χώρες μας, όπως για παράδειγμα στην Ουγγαρία. Γι' αυτό ε, Αυτά από την πλευρά της κυρίας Γιακονσάρη και ο, κύρι, ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. <clears throat> Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, την Σάντρα, για το εξαιρετικό της έργο, που συνοψίζει πάρα πολύ καλά τις σχέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία. Όλοι το γνωρίζαμε ότι οι σχέσεις μας με την χώρα αυτή δεν είναι οι καλύτερες δυνατόν, παρόλο που έχουμε δώσει πολλά. Ε, δύσκολα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον Πούτιν λέγοντας ότι αποτελεί έναν εταίρο της Ευρώπης. Ακούσαμε στην διάσκεψη των G20 στην Αργεντινή τον πρόεδρο Πούτιν θα συνεχίσει τον πόλεμο στα ανατολικά της Ουκρανίας. Όσο οι αρχές της Ουκρανίας παραμένουν στην εξουσία. Έτσι είπε, ήταν ξεκάθαρο αυτό που είπε και αντικατοπτρίζει πολλά και ξέρει και την επιθυμία της Ρωσίας να συνεχίσει να λειτουργεί μεροληπτικά παρά τις εκκλήσεις από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση πραγμάτων και ε, παρά ε, την κατάσταση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μια συνεργασία ακόμα και αν αυτή είναι αδύναμη, γιατί ο διάλογος αποτελεί ε, βασικό στοιχείο των αρχών μας. Η Ρωσία όμως δύσκολα τον δέχεται αυτό το διάλογο. Οπότε χαίρομαι που ζητάμε με την έκθεση αυτή μια νέα μορφή συνεργασίας με τη Ρωσία, εκεί όπου είναι αναγκαίο και εκεί όπου έχουμε ένα κοινό συμφέρον και επίσης ε, μιλάει και για μια επιλεκτική στάση απέναντι στα ενεργειακά, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος κτλ. Μην ξεχνάμε όμως ότι η Ρωσία δεν είναι μόνο ο Πούτιν, είναι και ο ρωσικός λαός. Και το λέω αυτό γιατί πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μας να διατηρήσουμε διάβολους επικοινωνίας με την κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να τους βοηθήσουμε εκείνους που αγωνίζονται για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, η επαφή με τον κόσμο είναι βασική. Πρέπει να την αθαρρύνουμε και να συνεχίσουμε. Και να συνεχίσουμε να συναντιόμαστε με τους ακτιβιστές, με τους δημοσιογράφους των ανεξάρτητων μέσων. Και τελειώνω με το κέντρο Memorial για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταδικάζουμε τη στάση της Τουρκίας απέναντι στην Ουκρανία, τη Γεωργία, ακόμα και την Μολδαβία. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας. Επόμενος, ο κύριος Αστροβίτσιος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ, συνάδελφοι. Συγχαρητήρια στην Σάντρα Καλνιέτε για το σχέδιο έκθεσής της που μας παρουσίασε σήμερα. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Και βλέπω πολύ καλό περιεχόμενο. Και ένα καλό μήνυμα. Στο τέλος της θητείας αυτής, δηλαδή το Κοινοβούλιο με την έκθεση αυτή συνοψίζει το έργο του και παρουσιάζει την πολιτική εικόνα όσον αφορά τις σχέσεις μας με τη χώρα αυτή. Πρέπει να ομολογήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι ότι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας ε, έπεσαν πολύ. Ξεκινήσαμε από το επίπεδο της στρατηγικής σχέσης με φιλοδοξία δεν αξιολογήθηκαν καλά. Ήταν περισσότερο μια ευχή, μια επιθυμία παρά μια κατάσταση πραγμάτων. Και φτάσαμε στον αντίποδα που πολλές φορές πρόκειται για προκλήσεις που δεχόμαστε από τη ρωσική πλευρά σε σχέση με οτιδήποτε προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του διεθνούς δικαίου, μετά από διάλογο και συνεννόηση με τους γείτονε. Εδώ βέβαια δεν τελειώνει η ιστορία. Οι ρωσικές δράσεις εξελίσσονται. Υπάρχουν ε, οι δραστηριότητες παραπληροφόρησης, κάτι το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο. Αυτά που γίνονται δηλαδή στα μέσα ενημέρωσης, στις κοινωνικές πλατφόρμες. Είναι ένας ανοιχτός πόλεμος κατά των ευρωπαϊκών αξιών και της αντικειμενικής πληροφόρησης. Εμείς πρέπει να προλαβαίνουμε τις δράσεις αυτές όμως. Θέλω να τονίσω ένα πράγμα στην έκθεση αυτή και γενικά όσον αφορά την κοινή μας θέση απέναντι στην πράξη Μακνίσκη όπως την ονομάζουμε για την Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει ένα καλό μηχανισμό για να τιμωρούμε και να επιβάλλουμε κυρώσεις. Πρόεδρε, τέλη Δεκεμβρίου οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών Υποθέσεων θα συναντηθούν για να συζητήσουν την Ολλανδική πρόταση που έχει να κάνει ακριβώς με αυτήν την πράξη και ζητώ από τους υπουργούς μας να διατηρήσουν τον τίτλο Μακνίσκι Act γιατί σημαίνει πολλά είναι κάποιος, ο Μακνίσκι, που σκοτώθηκε ακριβώς επειδή αγωνίστηκε κατά της διαφθοράς στο ρωσικό καθεστώς, στα υψηλότερα επίπεδα. Οι τέσσερις αυτές χώρες λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εγκρίνει την πράξη αυτή, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Εστονία, η Λετωνία και η Λιθουανία, πρέπει να αποτελέσουν ένα καλό παράδειγμα για τους υπόλοιπους, να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και να εγκρίνουν αυτή την πράξη Μαγνίσκη για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Στροβίσιους. Ολοκληρώνεται λοιπόν με τον τρόπο αυτό η συζήτηση για την ε, έκθεση για τις σχέσεις ε, Ρωσίας Ηνωμένων Πολιτειών, συγγνώμη, Ευρωπαϊκής Ένωσης, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 10 Ιανουαρίου 2019 στις 11 το πρωί. Επόμενο σημείο, ε, κυρίες και κύριοι, είναι η απαλλαγή του 2017 για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Μούντι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω εξ ονόματος της Ενίνα Γκίλ που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα. Ε, θα παρουσιάσω τη γνωμοδότηση της ΑΦΕΤΕ για την απαλλαγή 2017 όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η Νίνα λοιπόν αναφέρει ε, ορισμένα σημεία. Πρώτον υπογραμμίζει την ε, σημασία της εξωτερικής ε, πολιτικής και καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συνεχίσει να επενδύει στη στρατηγική επικοινωνία. Δεύτερον, υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η χρηστή οικονομική διαχείριση των αποστολών παρατήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Κομισιόν να σκεφτούν τον τρόπο με τον οποίο ε, ε, θα βελτιωθεί, να συντονιστούν έτσι ώστε να βελτιώσουν τις προσφορές των προμηθειών των εξωτερικών ε, συνεργατών. Επίσης, ε, επόμενο σημείο, ε, να ε, διασφαλιστεί περισσότερο και να εγγυηθεί περισσότερο η ασφάλεια των ατόμων που συμμετέχουν στις εξωτερικές αποστολές. Τέλος, να υπάρχει ισορροπημένη αντιμετώπιση των φύλων, κυρίως όσον αφορά σε ενδιάμεσο ε, ε, ε, επίπεδο διαχείρισης. Τέλος, η Νίνα εκφράζει την ικανοποίησή της γιατί το ποσοστό λάθους δεν είναι πάρα πολύ ψηλό, ωστόσο έχει ελαφρώς ε, μεγαλώσεις προς το τέλος του χρόνου και καλεί λοιπόν την ε, υπηρεσία να το λάβει υπόψη της. Ε, επίσης θεωρεί η Νίνα Γκίλε ότι το πρόγραμμα Global Europe είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, υποστηρίζει πλήρως τις στάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου όσον αφορά τις δαπάνες υπό το Global Europe και καλεί επιγόντως να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις αυτές. Επίσης, χρηστεί διαχείριση όσον αφορά τις αποστολές ε, των ε, παρατηρήσεων, παρατηρήσεων εκλογών ή στις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέταρτον, θεωρεί ότι δεν υπάρχει αρκετή ορατότητα ε, των, ε, της παρουσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλά ε, προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από αυτήν. Τέλος, όσον αφορά το τελευταίο σημείο για την απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υποστηριχτούν οι μεταρρυθμίσεις σε την Τουρκία. Θα πρέπει να δοθούν κονδύλια στην κοινωνία των πολιτών με έλεγχο της διαχείρισης. Τέλος, ε, όλες ε, οι ε, συστάσεις που έχουν γίνει από το ελεγκτικό συνέδριο και για την διαχείριση των κονδυλίων και τη μετανάστευση θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με τις τουρκικές αρχές για το τα ε, αυτά. Ε, τώρα, εάν έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις, ε, είναι εδώ ο, ο βοηθός της Νίνα Γκίλ και ίσως θα μπορούσε να σας απαντήσει. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 11 Δεκεμβρίου ε, τρέχοντος έτους στις 11 το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρους της. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μούντι. Ο κύριος Πρέντα από το ΕΛΚ. Αλλά σας υπενθυμίζω ότι πραγματικά έχουμε αργήσει πολύ δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ε, ε, ευτυχώς αυτή τη φορά δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό. Θα κάνω και εγώ σχόλια για τις δύο απαλλαγές, μια και παρουσιάστηκαν και οι δύο απαλλαγές. Όπως είπε και η ύπατη εκπρόσωπο στην Επιτροπή Οικονομικών, στα πλαίσια αυτών των, της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, ε, ληφθούν υπόψη και να εφαρμοστούν οι συστάσεις προηγούμενες και παρούσες ε, του ελεγκτικού συνεδρίου και οπωσδήποτε να υπάρχει σωστή και χρηστή διαχείριση των κονδυλίων σε γενικές γραμμές ε, είναι ε, θετικό, ε, θετική γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου και όσον αφορά τον διοικητικό προϋπολογισμό, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί χωρίς ιδιαίτερα λάθη. Να σας πω επίσης ότι πριν από δύο εβδομάδες οργάνωσα μια στρογγυλή τράπεζα με θέμα της ψευδής ειδήσει, παραπληροφόρηση κτλ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να το αντιμετωπίσουμε και με την απαραίτητη χρηματοδότηση. Είναι γεγονός ότι οι προβληματισμοί δεν είναι οι ίδιοι στην Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε και ακριβώς για να ε, αλλάξει η κατάσταση αυτή να δοθούν κονδύλια και να γίνει μια προσπάθεια όσον αφορά ε, τώρα ε, το ε, θέμα της ε, ισότητας των φύλων και αυτό είναι οπωσδήποτε ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει όσον αφορά την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως ε, και για την Ευρωπαϊκή Περισσοκή Εξωτερικής Δράσης, ε, είναι θετικό ε, το πόρισμα του ελεγκτικού συνεδρίου και επομένως θα πρέπει οι συστάσεις να ακολουθηθούν και να υλοποιηθούν. Υπάρχει ένα πρόβλημα βέβαια όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων που έχουν επιλεγεί. Θα πρέπει επομένως η ανάλυση να γίνει πιο στοχευμένη όσον αφορά την ΙΠΑ EPA ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη συνεχής αναφορά στο θέμα αυτό ε, στο, στο πόρισμα του ελεγκτικού ε, συνεδρίου και οπωσδήποτε διοικητικά να παρακολουθούμε τις χώρες αποδέκτες. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να βελτιώσουν τις διοικητικές τους ικανότητες και οι χώρες αποδέκτες. Πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να είναι πιο ε, αυστηρή όταν ελέγχει τους, τις προϋποθέσεις και τους όρους. Όσον αφορά τον εξορθολογισμό και την βελτίωση ε, των, ε, της οικονομικής διαχείρισης των παρατηρήσεων των εκλογών, πρέπει να πω ότι και οι δύο, τα δύο όργανα και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει από κοινού να διοργανώνονται και να συντονίζονται έτσι ώστε ε, οπωσδήποτε να βελτιωθεί η κατάσταση. Επίσης ε, ε, το θέμα των μεταναστών προσφύγων στην Τουρκία καθώς επίση και η βοήθεια στον Ήγερα και στο Μαλί για το ίδιο θέμα είναι σημεία πάρα πολύ σημαντικά τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν και τα αναφέρει άλλωστε και το πόρισμα του ελεγκτικού συνεδρίου. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Βίστησεν. Θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορο. Θέλω να ευχαριστήσω την, την εισηγήτρια. Θα υποβάλουμε τροπολογίες για τέσσερα θέματα. Πρώτον, για τι ε, αποστολέ παρακολούθηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που θεωρούμε ότι πρέπει να, υπάρχει καλύτερη διαχείριση σε αυτέ. Θέλουμε καλύτερη, πιο ενισχυμένη αναφορά στο ρόλο των κρατών μελών, καθώ είναι ε, εκείνοι που ηγούνται της ε, χάραξης εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θεωρούμε ότι αυτή η Task Force θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ε, κουτί της Πανδώρας, γιατί έχουμε και άλλους όρους εκπροσώπης, όπως για παράδειγμα γεωγραφικούς, και γι' αυτό είναι δύσκολο να διαχειριστεί, να, να διαχειριστεί κανείς όλα αυτά. Και ε, τέλος, υπάρχει το ζήτημα της Τουρκίας και του Ταμείου και της βοήθειας. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεργαστούμε με τη συγκίτρια. Ελπίζουμε να βρούμε συμβιβασμού. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βίστη. Θέλω και εγώ να σα να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία είναι η 11η Δεκεμβρίου. Πολύ σύντομα για την απαλλαγή 2017. Θέλω να αναφερθώ σε μια διάσταση Ακούστηκε και μια κάπως επικριτική παρατήρηση από την, πλευρά, από την πλευρά της ε, Νίνα Γκίλ για τους εκλογικούς παρατηρητές. Εκεί ε, υπάρχει μια αναφορά σε χρηστή οικονομική διαχείριση κτλ. κτλ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εκφράζουμε την υποστήριξή μας στην ε, διαδικασία που έχει ακολουθηθεί μέχρι στιγμής, διότι εξασφαλίζει ταχύτητα και αποτελεσματικότητα λαμβανομένων υπόψη και των περιστάσεων που επικρατούν πολύ συχνά επί τόπου. Κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι τα χρήματα είναι πολλά. Όμως πρέπει να ξέρετε για παράδειγμα στο Πακιστάν πρέπει κανείς για να μετακινηθεί να ε, νοικιάσει θωρακισμένα οχήματα για να μπορεί να μετακινηθεί μέσα στη χώρα. Το να Στέλνουμε λοιπόν εκλογικούς παρατηρητές, είναι σημαντικό, είναι τόσο σημαντικό ώστε δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψη έτσι μονοδιάστατα η οικονομική πτυχή του θέματος. Έχει πολιτική σημασία. Γι' αυτό και θα έλεγα να κρατήσουμε ε, στο επίκεντρο της προσοχής μας το πραγματικά σημαντικό και όχι το δευτερεύον. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Με αυτό ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενο θέμα. Ανάπτυξη της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση. Η συγγήτρια είναι η κυρία Σωράγια Πόστ. Αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα και αργότερα. Δεν έχουμε τώρα πολύ ώρα, γι' αυτό Σωράγια, σε παρακαλώ, όσο πιο σύντομα γίνεται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν είναι και εύκολο αυτό που μου αναθέτεται. Θα προσπαθήσω. Πρώτον, χαίρομαι που μπορώ να σας παρουσιάσω αυτό το σχέδιο έκθεσης για την ανάπτυξη ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση. Βλέποντα τον κόσμο σήμερα, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι η πρόληψη συγκρούσεων και η διαμεσολάβηση είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα πρέπει απλώς να προωθηθεί αλλά και να ενισχύσει το επίπεδο των εργασιών της στον τομέα αυτών. Η πρόληψη συγκρούσεων ε, είναι ε, τμήμα ε, του, του, του, του πυρήνα αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργήθηκε γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέσο για την πρόληψη συγκρούσεων, ως εγχείρημα ειρήνης. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει τις ικανότητες της σε αυτόν τον τομέα στην πρόληψη της, των συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση. Η έκθεση λοιπόν επικεντρώνεται στο πώς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να είναι πιο ισχυρά και να έχουν πιο συνεπή στάση όσον αφορά την πρόληψη και τη διαμεσολάβηση. Στη διαδικασία αυτή ε, έχουμε λάβει δηλώσεις από όλους τους εμπλεκόμενους ότι χρειάζεται να εμπλακούμε πολύ περισσότερο και να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας στους τομείς αυτούς. Επίσης, Πολύ σημαντικό είναι το, το θεματολόγιο του ΟΗΕ για την ε, ειρήνη και την ασφάλεια, ώστε να ενισχυθεί η, ε, η δημοκρατική λήψη αποφάσεων, η ισότητα των ε, φύλων και η εξασφάλιση της μιας βιώσιμης ειρήνης και ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει βεβαίως τις συμφωνίες αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον κόσμο ως βασικός διαμεσολαβητής και συνεισφέρον σε διεθνούς οργανισμούς και μέσα ε, χρηματοδότησης. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα αυτά ε, συνοδεύονται από μεγαλύτερη ευθύνη για την ανάληψη δράσεων για την ειρήνη και την προώθηση τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη για όλου του ανθρώπου. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα, τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης με καλύτερο τρόπο γιατί αυτοί συνεισφέρουν σημαντικά στο έργο για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση. Πρέπει επίσης να ενισχύσουμε ε, τις ε, δεσμεύσεις μας και την προσήλωσή μας και χαίρομαι που κάτι τέτοιο έχει επιδείξει και αποδείξει με την στάση της και η πατή εκπρόσωπος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης ε, διαδραματίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στην ε, κοινοβουλευτική διπλωματία. Και αυτό είναι θετικό. Σε όλες τις εργασίες πρόληψης συγκρούσεων είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας πάντοτε τις γυναίκες που είναι τα μεγαλύτερα θύματα των συγκρούσεων και είναι και εκείνοι που ε, συνήθως αποκλείονται από, την, ε, ε, από τις εργασίες και τις διαδικασίες πρόληψης. Αυτό δεν είναι λογικό και υπονομεύει άμεσα την επιτυχία των εργασιών συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και κάνω ρητή έκκληση για τις γυναίκες, ώστε αυτές να εκπροσωπούνται πάντοτε σε όλα τα στάδια των εργασιών πρόληψης συγκρούσεων και την ενίσχυση των σχετικών προσπαθειών. Επίσης, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χαράξει μακροπρόθεσμες προτεραιότητε και στρατηγικές και να αναπτύξει μια ε, συνεπή ε, και συνεκτική αρχιτεκτονική. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα. Και κάνω τις, τις εξής στην κατεύθυνση αυτή. Πρέπει να δημιουργηθεί ε, ένα ε, ενωσιακό υψηλού επίπεδου συμβούλιο για τη διαμεσολάβηση που θα βοηθήσει την ενίσχυση αρχών όπως είναι ε, η ισότητα των φύλων, κάτι που θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκρίνεται σε προκλήσεις έγκαιρα. Επίσης, θέλω να θεσπιστεί θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέσβη για την ειρήνη που ε, θα αποδείξει και την βούλησή μας να ενισχύσουμε αυτή τη διάσταση των εργασιών μας. Επίσης, καλό να δημιουργηθεί ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρέπει να αναπτύξει περιττέρω τις υπηρεσίες πρόληψης συγκρούσεών της, καθώς και τις ικανότητες της στα ζητήματα ισότητας των φύλων ε, και συγκρούσεων. Και πρέπει επίσης να υπάρξουν επενδύσεις στον τομέα αυτό μαζί με την ε, διάδοση και την ανταλλαγή γνώσεων. Οι γνώσει στον τομέα τη πρόληψη συγκρούσεων και διαμεσολάβηση θα πρέπει να είναι κοινό κτήμα όλων των θεσμικών οργάνων. Η υπηρεσία εξωτερική δράση χρειάζεται επίση αναλύσει ε, όπου θα λαμβάνουν υπόψη τους την διάσταση του φύλου. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα βαθύνουμε τις συγκρούσεις λόγω έλλειψης γνώσεων και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η διάσταση του φύλου λαμβάνεται πάντοτε υπόψη στο έργο της πρόληψης. Πρέπει να, να αντιμετωπίσουμε τις γενεσιουργές αιτίες των συγκρούσεων και να ενισχύσουμε την ε, βιώσιμη ανάπτυξη για να αντιμετωπιστούν αυτές οι αιτίες Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε προσοχή μας στη, στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη, τη δικαστική μεταρρύθμιση, το κράτος δικαίου και αυτό θα πρέπει να είναι μια διαδικασία που θα περιλαμβάνει και την κοινωνία των πολιτών και τα προγράμματα φύλου. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές διαστάσεις των εργασιών μας για την πρόληψη συγκρούσεων και πρέπει ε, όλες οι, οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει μ, μεγάλη σημασία ε, στην πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή της έχει αποδείξει ότι η διπλωματία και η διαμεσολάβηση μπορούν να αποφέρουν αποτελέσματα ακόμα και στις πιο δύσκολες διεθνείς καταστάσεις. Μία, ένα λεπτό ακόμη θέλω, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό ακόμη. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντικό να βασιστούμε στις επιτυχημένες δραστηριότητες και τα επιτεύγματα που έχουμε ήδη ε, στην πορεία μας. Πρέπει να ενισχύσουμε το συντονισμό μεταξύ των ε, δραστηριοτήτων και των δράσεων μας και εδώ προτείνω η Αντιπρόεδρος να είναι ε, υπεύθυνη για το συντονισμό των εργασιών και των ε, δράσεων διαμισολάβησης μας και να διευκολύνει τον διάλογο και τις σχετικές μας δραστηριότητες. Ο κύριος Πρόεδρος, κυρία Πόστ, έχετε μιλήσει ήδη 7 λεπτά. Τέλος, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κατευθύνει επαρκείς πόρους και να προβλέπει προπολογισμό ώστε αυτέ οι πολιτικέ μα φιλοδοξίε να μπορούν να μετουσιωθούν σε πράξη. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να υπάρχει ειδική γραμμή του προπολογισμού για τη διάσταση του φύλου και για το, για το επαρκές προσωπικό που χρειάζεται όλα αυτά που ε, προβλέπουμε ότι πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω συνεργασία με τους Κιώδης. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πρέντε υποσχέθηκε ότι θα είναι πάρα πολύ σύντομο Για να δούμε. Ναι, όπω πάντα, Πρόεδρε. Για τον συνάδελφο Ντανζόν, που δυστυχώ δεν είναι εδώ, θέλω να μιλήσω. Ο στόχο της έκθεσης αυτής είναι να προτείνει συστάσεις για την δημοσιονομική ικανότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Αξίζει τον κόπο, το κείμενο παρουσιάζει ε, ιδιαίτερε και ενδιαφέρουσε ιδέε για την διαμεσολάβηση. όμω λέει ο ε, αμφιβάλλω για την προστιθέμενη αξία της έκθεσης αυτής όσον αφορά τους τύπους αλλά και την ουσία. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο το κατάλληλο είναι μια τέτοια έκθεση και επί της ουσίας είναι προβληματικό το κείμενο. Μιλάει για την επίλυση σε βάση του φύλου με ανάλυση που βασίζεται κάθε φορά στο φύλλο και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση βάσει αυτού να αντιμετωπίσει τις συγκρούσεις, κάτι το οποίο περιορίζει πάρα πολύ το θέμα. Εξού και θα υποβάλω τροπολογίες που να εξισορροπούν το κείμενο, λέει ο κύριος Δαζό. Ευχαριστούμε κύριε Πριντά. ο κύριο Κούκαν τώρα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ξέρω από θέματα διαμεσολάβησης και γι' αυτό έχω να πω κάτι. Δυστυχώς έχασα την παρουσίαση της κυρίας Πόστ αλλά σε ένα λεπτό θέλω να πω ότι είναι πολύ καλό που συζητάμε αυτό το ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό που ετοιμάζουμε έκθεση. Και από τη δικιά μου εμπειρία σε συγκρούσεις όπως αυτές στην γειτονία μας ή στα Δυτικά Βαλκάνια, χρειάζεται πολιτική δέσμευση με διαμεσολάβηση και για την πρόληψη κρίσεων. Χαίρομαι λοιπόν για το σχέδιο αυτό έκθεσης που θέτει ένα σαφές πλαίσιο προκειμένου να διορθωθεί καλύτερα η πολιτική αυτή πρόθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι θα έχει τις κατάλληλες ικανότητες για να προβεί σε δράση. Θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες που θα αναφέρονται σε αυτά και βέβαια με το συνήθι διάλογο που χρησιμοποιούμε και στην περίπτωση της Μακεδονίας. Λέει ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κούκαν, λέει ο πρόεδρος, και σας ευχαριστώ όλους. Κύριε Πώς, θέλετε να αντιδράσετε πραγματικά 30 δευτερόλεπτα σας δίνω. Όχι, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Απλώς προσβλέπω κι εγώ στην ετοιμασία αυτή της έκθεσης. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε καλά μαζί. Πρόεδρος, υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 10η Δεκεμβρίου. Ερχόμαστε στο... 10η Ιανουαρίου, 10η Ιανουαρίου. Ερχόμαστε στο επόμενο θέμα. Πρόκειται για την ε, κοινή συνεδρίαση που έχουμε την Επιτροπή Ανάπτυξη για τη θέσπιση μηχανισμού γειτονία, ανάπτυξη και διεθνού συνεργασία. Βάσει τη διαδικασία που από κοινού επιτροπέ εκπονούν ε, έκθεση, ε, ετοιμάζουμε από κοινού την έκθεση αυτή και θα καταλήξουμε σε κοινή συνεδρίαση στις 4 Φεβρουαρίου. Είναι μια σημαντική διαδικασία γιατί έτσι θα καθορίσουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τρίτες χώρες με 90 δισεκατομμύρια περίπου από το 2021 μέχρι το 2022. που θα αποτελέσουν και τη βάση για τη σημερινή μας συζήτηση. Έχουμε λίγο χρόνο, οπότε θα δώσω το λόγο αυτή αμέσως στην πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξη, την Λίντα Μακάβιν, για τα εισαγωγικά της σχόλια. Ναι, ευχαριστώ. Το μόνο που θέλω να